όχι αρέντολοι, η επιβεβαιώνεται. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζήτησε να αναλάβει ο κύριος Σέργιο Γκουτιέρες την θέση της κυρίας Μαγδαλένα Αλβάρες Άρσα στην αντιπροσωπεία με τη Ρωσία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι, οπότε εγκρίνεται και αυτό. Έλαβα από το Συμβούλιο την θέση ε,